τον κύριο Μούρεσαν. Nous avons reçu... Ως μέλη της Επιτροπής Προβλογισμού, αλλά και ειδικέ επιτροπές ε, λάβαμε στις 2 Ιουλίου τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης ε, για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε αυτή την πρώτη αξιολόγηση εμπειρογνώμονές της. Μια προεκτίμηση. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Ιουρέλ για να μας τα παρουσιάσει αυτά. Αν και έχουμε την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, κατάλαβε καθόλου τι τη ζητάμε σε κάποιες περιπτώσεις. Και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Ντανιέλ Βιώτη, γενικό εισηγητή μας. Είστε έτοιμος κύριε Ιουρέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία σύντομη εισαγωγή. Στις 3 Μαΐου το Κοινοβούλιο μεταβίβασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναν κατάλογο 344 προκατακτικών προτάσεων για πολιτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικών δράσεων σημειώνουμε ότι από το 2016 και για τρία χρόνια συνεχόμενο ο αριθμός των προκαταρκτικών προτάσεων είναι πάνω από τον μέσο όρο των, 200 προτάσεων που λάβουμε τα προηγούμενα χρόνια. Λάβουμε 350 προτάσεις και Και αυτό απαιτεί μεγάλη Προσπάθεια σε διοικητικό επίπεδο από τις υπηρεσίες. Έχουμε αξιολογήσει όλες τις προκαταρκτικές προτάσεις εντό του ε, χρονικού περιθωρίου που μας δόθηκε και πέρα από αυτές τις 344 η αξιολόγηση τη επιτροπή είναι ότι 42 προτάσεις θα μπορέσουν να εφαρμοστούν όπως προτείνεται 26 ε, προγράμματα πιλωτικά. 56 προτάσεις μπορούν να εφαρμοστούν εν μέρη αν ανασχεδιαστούν οι υπό συγκεκριμένε ε, προποθέσει. Αυτά είναι στην κατηγορία Β. Υπάρχει και κατηγορία C. 84 προτάσεις οι οποίε καλύπτονται πλήρω από, από τρέχουσες ε, προτάσεις ή νομικές προϋποθέσεις και από ευρωπαϊκές δράσεις και η κατηγορία D στην οποία αξιολογήσαμε με 61 προτάσεις οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια για να εφαρμοστούν είτε λόγω ε, νομικής ασυμβατότητας είτε επειδή έχουν ήδη εφαρμοστεί στο παρελθόν. Είμαι έτοιμο να απαντήσω σε ερωτήματα. ξεκινήσατε λοιπόν τη συζήτηση για να πάρει ο κύριος Βιώτη το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Βρισκόμαστε σε μία φάση αρκετά ενδιαφέρουσα της προσπάθειας η οποία γίνεται για τις προπαρασκευαστικές και πιλωτικές δράσεις. Ο συμπαθής συνάδελφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγκαζόμαστε να συζητάμε όλα αυτά τα θέματα τα επιμέρους γιατί δεν έχουμε ιδιαίτερες νομοθετικές εξουσίες. Αν αποκτήσουμε επιπλέον νομοθετική εξουσία τότε θα ασχολούμεθα μόνο με τα γενικά και σημαντικά. Ευχαριστώ πάντως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσπάθεια την οποία έχει κάνει μέχρι τώρα. Είναι μια προσπάθεια η οποία μας επιτρέπει σε όλους να εμβαθύνουμε σε ένα θέμα το οποίο είναι θα έλεγα κυρίως πολιτικό και όχι μόνο τεχνικό. Θα ήθελα επίσης ε, να πω δύο πράγματα. Η αξιολόγηση την οποία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και την οποία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αμυγός ε, πολιτικού χαρακτήρα. Φυσικά και θα σεβαστούμε τις προτάσεις τις οποίες έχει κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά από την άλλη θα κάνουμε μία αξιολόγηση και εμείς στο εσωτερικό της Επιτροπής μας πολιτικού χαρακτήρα, υπενθυμίζοντας ότι τα πιλωτικά προγράμματα είναι ένα εξαιρετικό μέσο το οποίο έχει στη διάθεσή του το Κοινοβούλιο για να συμπληρώνει τις πολιτικές οι οποίες δεν καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να δίδονται επακριβέστερες απαντήσεις από ό,τι τα καταφέρνει ο προϋπολογισμός σε κάποιους τομείς. Όλα αυτά δεν είναι, βασί περιπτώσει, μικροπράγματα. Ε, ζητώ συγγνώμη από τους διευμηνείς γιατί το λέω με πολύ συγκεκριμένο τρόπο ε, δεν είναι και κάτι το οποίο αναφέρεται μόνο και αφορά αποκλειστικά τα μεμονωμένα κράτη-μέλη, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βρούμε ένα πακέτο ισορροπημένο το οποίο να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τις οποίες έχουν οι πολίτες και γι' αυτό ακριβώς και μετά από τις προσπάθειες τις οποίες έχει κάνει τον προηγούμενο χρόνο ο κύριος Μούρεσαν ε, σκοπεύω να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο με πιο ικανοποιητικό τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Βιώτη. Ε, κύριε Μούρεσαν, αν θέλετε μπορείτε να πάρετε το λόγο και να μεταφέρετε και τις δικές σας εμπειρίες για τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Δεν υπάρχει κάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τα πολιτικά προγράμματα που αναπτύσσουμε για το 2018 δεν υπάρχει κάτι να προσθεθεί από την πλευρά μου, αλλά αν ε, μου δώσετε το λόγο, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τον ενιαίο για τη στολή που φοράει ο συνάδελφος ο κύριος Ντεπρέ, βλέπω κόκκινο και κίτρινο και να πω δεν ξεχνάμε και τη Γαλλία κύριε Πρόεδρε δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο για τα πολιτικά προγράμματα από την πλευρά μου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 το ρόλο μας. Εφόσον κάθομαι σε αυτήν την πλευρά, έχω τη δυνατότητα να δείξω την προτίμησή μου. Εσεί όμω που στο πρώτο πρέπει να είστε ουδέτερο, και αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε εσά και σε μένα. Έχουμε διαφορετικό ρόλο. Δεν έχει να κάνει με το πόσο δυνατά είναι τα αισθήματά μα. Να εκφράσω τον κύριο Βιώτη για τα σχόλιά του. Θα ήθελα όμω να μοιραστώ και κάποιου προβληματισμού με εσά. Ξέρω ότι ανησυχείτε και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε ε, ομοφωνία, να έχουμε συνένεση ώστε να έχουμε μια πολιτική ισορροπία το οποίο θα πρέπει να αντικατοπτριστεί και στην επιλογή των προπαρασκευαστικών δράσεων και των πολιτικών προγραμμάτων. Ωστόσο, διστάζω. Δεν μου αρέσει να δεν συμφωνώ πλήρω με τον κύριο Βιώτη. Και αυτό έχει να κάνει με τις ελευθερίες που μπορούμε να έχουμε όσον αφορά την ε, ταξινόμηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλουμε να λάβουμε υπόψη τις δύο πρώτες κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ίσως αν συμφωνήσουμε να υπάρξουν εξαιρέσεις με την κατηγορία C. Όμως θεωρώ ακόμα ότι αυτό θα μπορούσε να είναι λίγο ε, περίεργο, λίγο δύσκολο αυτό όμω πράττω λίγο στου συναδελφού μου ότι ναι, έχετε πολιτικά προγράμματα, αλλά θα πρέπει να σα πω ότι η προτεραιότητα θα δοθεί στην κατηγορία C. Και αν συμφωνούμε και στην κατηγορία Β, B. Αλλά δεν μπορούμε να πραγματευτούμε με αυτού που έχουν πάρει κάποια καλύτερη κατάταξη. αν η Επιτροπή έχει κάνει τη δουλειά, δεν υπάρχει λόγος ε, να κάνουμε το ίδιο πράγμα δεύτερη φορά. Απλώς θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Αν θεωρούμε ότι υπάρχουν προβλήματα με τις αρμοδιότητες, θα, θα είναι δύσκολο να αποδεχτούμε αυτά τα πιλωτικά προγράμματα. Η πολιτική μου ομάδα Ευχαριστώ θα εμπλακεί σε αυτές τις συζητήσεις, όμως αυτή είναι η όρη που έχουμε θέσει και υπάρχουν κάποια όρια και σας έχω θέσει τα όρια, οπότε ελπίζω να μπορέσετε να το κάνετε. Ε, euh, στην περίπτωση που δεν υπάρξει κατανόηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει και εμείς να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Κύριε Σόλμπρεχτ, εγώ νομίζω παρουσίασα προγράμματα στην κατηγορία Α Συγχαρητήρια λέει ο πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει, έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε μία συζήτηση για την έννοια της προπαρασκευαστικής δράσης και της πιλωτικής δράσης. Το θέμα δεν είναι η διαφορετική κατηγορία α, β ή γ. Το θέμα είναι πώς θα οργανωθούμε και ποιος θα είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή, ποιος θα το κάνει αυτό. Η πραγματική ερώτηση είναι εξή Εμείς σαν παράδειγμα έχουμε τις πολιτικές ε, απόψεις που είναι σημαντικές για μας, τις στέλνουμε ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή είναι αυτή η οποία μας λέγει ότι κοιτάξτε ίσως το θέμα αυτό να είναι πολιτικό για σας αλλά δεν είναι εφικτό για μας. Και μάλιστα δεν είναι εφικτό γιατί δεν έχουμε ε, και το κατάλληλο προσωπικό. Θα πρέπει να οργανώσουμε διαγωνισμούς και δεν είναι και στις αρμοδιότητές μας και ό,τι άλλο θέλετε. Το θέμα δεν είναι ότι οι ιδέες μας θα καθορίσουν τον τρόπο οργάνωσης, αλλά οι ιδέες μας οι οποίες θα πρέπει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνουν πραγματικότητα. Εγώ είμαι εδώ και 14 χρόνια. Κάθε χρονιά τα ίδια έχουμε. Πώς μπορεί να κρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι σημαντικό. Αυτό είναι το πολιτικό θέμα. Αυτό το θέμα δεν είναι αυτό το οποίο που θεωρούμε σαν σημαντικό αν είναι ή δεν είναι σημαντικό. Το θέμα είναι ποιος το αποφασίζει. Συνεπώς λοιπόν δημιουργούνται συνεχώς ε, παρανοήσεις και γι' αυτό ακριβώς ε, τα πιο έμπειρα αν θέλετε ε, μέλη είναι αυτά τα οποία προσπαθούν να συνεννοηθούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν παρουσιάσουν την πρότασή τους. Γιατί θα μας πει η Επιτροπή αν είναι εφικτό ή όχι. Αν μας πει ότι δεν είναι εφικτό σταματάμε. Λοιπόν, δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Θα ήθελα επί τη βάση μιας εμπειρίας την οποία είχε πως ε, ε, αν πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάτι δεν είναι εφικτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι πράγματι εφικτό και θα πρέπει να δούμε και εμείς πώς ακριβώς στο εσωτερικό της Επιτροπής λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις. Πρόκειται δηλαδή για μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια. Κύριε Βιώτη, νομίζω ότι τα πράγματα είναι σαφή. Έχετε την υποστήριξη και του κυρίου Μουρεσάν. Σταματάμε με το θέμα αυτό, περνάμε στο επόμενο. Ε, τις προβλέψεις πληρωμών αποφασίστηκε να μην γίνει διοργανική συνάντηση για τις πληρωμές το μήνα Ιούλιο ε, για να αντικαταστήσουμε την συνεδρίαση αυτή θα μας παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τις προβλέψεις της για την εφαρμογή του προϋπολογισμού η οποία διανεμήθηκε χθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε στο νου μας και το προσχέδιο προϋπολογισμού του 19 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δίνω το λόγο επίσης πάντα στον κύριο Ιουρέλ, εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Budget. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να δώσω μια σύνοψη της κατάστασης εφαρμογής εκτέλεσης του προπολογισμού του 2018 ε, σε πιστός πληρωμών. Αυτό είναι το θέμα της ανταλλαγής απόψεων σήμερα. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, έχουμε διανύμει την έκθεση παρακολούθησης και πρόβλεψης και θεωρώ ότι εν συντομία μπορώ να πω ότι η εκτέλεση ως στιγμή είναι αρκετά θετική. Στις 30 Ιουνίου εκτελέσαμε πληρωμές άνω των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορά το 56-57% των διαθέσιμων ε, πιστώσεων πληρωμών. Αν το συγκρίνουμε αυτό με την ε, ημέρα εκτέλεση ε, πέρσι βλέπουμε ότι είναι υψηλότερο το ποσοστό και σε ε, αριθμούς κατά 10 δισεκατομμύρια και κατά 7 με 8% πάνω. Επίσης, έχουμε, είμαστε μπροστά από το πρόγραμμα σε σχέση με τις προβλέψεις για φέτος που και αυτές αποτελούν κομμάτι της έκθεσης η οποία διανεμήθηκε χθε. Και αυτό ισχύει για όλα τα headings, εκτός από το 4, όπου υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση σε σχέση με τις προβλέψεις, του τίτλους. Θα μπορέσουμε όμως να συμβαδίσουμε πριν το τέλος του χρόνου. Θα δώσω μια σύντομη σύνοψη ανατίτλου, ξεκινώντας από τον τίτλο 1α. Η εκτέλεση βρίσκεται στο 50% που είναι περισσότερο από την ίδια ε, εποχή πέρσι, που είναι 45% 10 εκατομμύρια, υπό εκατομμύρια τον, δισεκατομμύρια υπό αυτόν τον τίτλο. Είμαστε πιο πάνω από τις προβλέψεις για τις 30 Ιουνίου αυτού του έτους. Είμαστε στο 49% και οι προβλήψεις ήταν στο 46%. Πολύ σημαντικό επίσης είναι και ο ρυθμός ε, εκτέλεσης για τον τίτλο 1B, συνοχή, που στις 30 Ιουνίου έφτασε στο 39,2%. Βρισκόμαστε μπροστά ελαφρώς από τις προβλέψεις για την 20 και είναι αρκετά πιο υψηλό από ό,τι στις 30, ήταν στις 30 Ιουνίου πέρσι και σε σχετικούς όρους. Είμαστε 5 ε, δισεκατομμύρια πιο πάνω και 9% πιο πάνω ως ποσοστό εκτέλεση σχέση με το 2017. Υπό τον τίτλο 1β η Επιτροπή έχει πληρώσει 18 δισεκατομμύρια 16,5 η μεγάλη η πλειοψηφία αφορά τη νέα γενιά προγραμμάτων για το 2014 και 2020 και τα υπόλοιπα αφορούσαν τα πράγματα του 2007-2013. Πάμε στον τίτλο 2. Ε, το Ταμείο Εγγύσεων για τη Γεωργία, έχει εκτελέσει 48%, 47 δισεκατομμύρια, επίσης 84% Όσον αφορά τα άλλα προγράμματα, υπό τον τίτλο 2, βλέπουμε μια παρόμοια πρόοδο στην εκτέλεση. Έχουμε εκτελέσει 57%, 7,5 δισεκατομμύριο για τα υπόλοιπα προγράμματα εκτός από το EGF και εδώ είμαστε πιο μπροστά από τις προβλέψεις. Το 2017 είμαστε στο 50%, άρα μπορώ να πω ότι έχουμε, είμαστε πολύ ψηλά στην εκτέλεση στον ε, τίτλο 2, στον τίτλο 3. Είμαστε στο 48%, 1,4 δισεκατομμύρια, σχετικά υψηλότερα από την πρόβλεψη, αρκετά πιο ψηλά από την ίδια περίοδο του περασμένου έτους. Όπως είπα, στον τίτλο 4 είναι ο μόνος τίτλος στον οποίο έχουμε καθυστερήσεις. Έχουμε εκτελέσει 3,2 ε, δισεκατομμύρια σε πληρωμές, που είναι μονάχα το 34% του τίτλου και η πρόβλεψη ήταν 3,9 δισεκατομμύρια. Άρα είμαστε 0,7 δισεκατομμύρια πίσω σε σχέση με πέρσι. Πέρσι είμαστε στο 3,8 δισεκατομμυρία, οπότε και εδώ έχουμε καθυστέρηση. Τίτλος 5. Εδώ η εκτέλεση δεν ε, μας εκπλήσει, είμαστε στο ίδιο επίπεδο με την πρόβλεψη και με τα επίπεδα του περασμένου έτους. Έχουμε εκτελέσει το 48% των πληρωμών. Όσον αφορά το δεύτερο μισό, το δεύτερο εξάμεινο, το μισό του έτους, τα νέα επόμενα σημαντικά στοιχεία θα είναι η υποβολή των ε, επικαιροποιημένων ε, προβλέψεων των κρατών μελών για τη συνοχή που τα περιμένουμε στο τέλος του μήνα, τα οποία θα τα αναλύσουμε και θα εξάγουμε συμπεράσματα. Όπως και σε προηγούμενα έτη, οι προβλέψεις είχαν μεγάλη συγκέντρωση πληρωμών τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο και συγκεκριμένα για τον τίτλο 1B. Άρα θα αξιολογήσουμε αυτές τις προβλέψεις των κρατών μελών κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και στις αρχές του Σεπτεμβρίου και σε παράλληλα Επιτροπή κάνει την ε, ετήσια άσκηση μεταφορών η οποία θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο και από κοινού η αξιολογήση των κρατών μελών και η έκθεση της Επιτροπής θα μας δείξει, κατα, ε, δείξει σε τι επίπεδο βρισκόμαστε όσον αφορά τον Global Transfer. Αυτή τη στιγμή έχουμε εντοπίσει στην πρόβλεψη μία έλλειψη πιστώσεων πληρωμών υπό τον τίτλο 1α κατά 240 εκατομμύρια και αφορά τα προγράμματα ITER Erasmus Plus και πυρηνική ασφάλεια. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο και αναμένουμε ότι στο πλαίσιο του Global Transfer θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις ελλείψεις στον τίτλο 1α ε, με μεταφορές από άλλους ε, τίτλους. Θα σας υποβάλουμε προτάσεις ε, σχετικές. Σε αυτή τη φάση, λοιπόν, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ε, ελλείψεων στις ε, πληρωμές. Αναμένει πλήρη εκτέλεση του προπολογισμού και ελπίζω να μην χρειαστεί να, έχουμε τέτοια επεισόδια με πέρσι και να μπορέσουμε ε, να σας παρουσιάσουμε ένα προπολογισμό με μείωση των πιστώσεων πληρωμών, αλλά όπως είπα, το βασικό στοιχείο θα πρέπει να μας ε, δώσει, ε, να μας παρέχει κάποια εμπιστοσύνη θα είναι το σε εκθέσεις αξιολόγησης των κρατών μελών. Αυτή είναι η γενική εικόνα και είμαι διαθέσιμος ε, για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Ουραλ. Σας ευχαριστώ. Στην παρούσα φάση θα δώσω το λόγο στον κύριο Μούρη σαν γενικό εισηγητή γιατί πρόκειται για πληρωμές ε, που αφορούν το οικονομικό έτος 2018. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά οι προβλέψεις για τις πληρωμές φαίνονται πιο ενθαρρυντικές από ότι τα περασμένα έτη. Έχει απορροφηθεί η καθυστέρηση και τα προγράμματα επιτέλους έχουν αρχίσει να φτάνουν σε μια ταχύτητα λειτουργίας κανονικής και σε πραγματικού, σε απόλυτες τιμές μάλλον και σε σχετικές υπάρχει μια σημαντική αύξηση και αυτό είναι αξιοσημείωτο όσο και θετικό. Τώρα, Επίσης καλό ήταν που η γενική εικόνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της αξιολογήσεις της ήταν ότι είναι επαρκείς οι πόροι που έχουν προγραμματιστεί για τις πιστώσεις πληρωμών για φέτος. Αλλά Ταυτόχρονα από την άλλη βλέπουμε ότι οι προβλέψεις είναι λίγο χαμηλότερες στην κατηγορία, στον τίτλο 1α και 1β. Και τι σημαίνει αυτό. Ότι οι προβλέψεις των κρατών μελών τείνουν να είναι όλο και πιο ακριβής. Δηλαδή τα κράτη-μέλη δεν υπερεκτιμούν τις δυνατότητες απορρόφησης που έχουν. Ε, ε, τώρα στην αρχή της επταετούς πραγματικής περίοδου. Αυτό το παρατηρεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι χρειαζόμαστε το επόμενο διάστημα μέχρι το τέλος του PDP θα πρέπει να έχουμε τις προβλέψεις των κρατών μελών ως αξιόπιστα στοιχεία. Γιατί τον τίτλο 2 θέλω κάτι να ρωτήσω. Βλέπω σημαντική απόκληση από τις προβλέψεις. 37 δις ε, ε, αξιώσεις πληρωμών και 32,7 είναι οι προβλέψεις. Πολύ ψηλότερο από την ε, απορρόφηση πέρυσι που ήταν 33 δις. Τώρα είμαστε στο 85% απορρόφηση σε σχέση με 75% πέρυσι τέτοιο καιρό. Θα ήθελα να μάθω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς έγινε αυτό, πώς προέκυψε αυτή η διαφορά. Η πιστός πληρωμών δηλαδή που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για φέτος είναι επαρκής. Αυτή ήταν μια ερώτηση για το τίτλο 2 και δεν έχω τίποτα περισσότερο προς στιγμή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αμέσως στη συνέχεια κύριος Βιώτη για τον προϋπολογισμό του 2019. Α, βγήκε. Έφυγε ο κύριος Βιώτη. Δεν ξέρω, συνάδελφοι, ποιοι θέλετε από να πάρετε το λόγο. Κανείς. Κάτι να πω μόνο. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι η ε, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ε, δεν ε, είχε παρκή απορρόφηση. Τώρα βλέπω ότι είναι στο 79,5% απορρόφηση των πληρωμών. Τι έγινε. Επιτέλους πήρε μπρος αυτή η διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και για το Εράσμος. 68% ε, απορρόφηση των πληρωμών. Αυτά τα δύο στοιχεία θα μπορούσαν να δώσουν έτσι μεγάλα επιχειρήματα ε, στο Γενικό Εισήγητη για την ε, κατάρτιση του προεπλεγισμού του 2019. Αφού δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, κύριε Ουρέλη, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για να απαντήσω σύντομα στην ερώτηση του κύριου Μουρεσάν. Είναι φυσιολογικό αυτό το φαινόμενο, το παρατηρούμε ετησίως στην κατηγορία στον τίτλο 2 και ιδιαίτερα ε, για το Ταμείο Εγγυήσεων για τη Γεωργία. Ε, ο κύριος όγκος των πληρωμών απορροφώντας στην αρχή του έτους φέτος η κατάσταση που διαπιστώνουμε είναι μάλλον επιστροφή στην κανονική ταχύτητα απορρόφησης από ότι ε, τα έτη 2016 και 2017 που ήταν μάλλον βραδία η εκκίνηση. Το 85% λοιπόν που παρατηρούμε είναι το φυσιολογικό και μπορώ να το επιβεβαιώσω απαντώντας στην ερώτησή σας ότι δεν πρόκειται ε, φέτος να υπάρξει πρόβλημα στην απορρόφηση των κονδυλίων για τη γεωργία. Ευχαριστώ. Voilà, απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις που σας ε, τέθησα. Για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Το 2020 μήπως ε, μείνουμε από πιστώσεις. Έλεγα ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων που υπάρχει πολύ μεγάλη απορρόφηση. 79,5%. Και μετά από τις αποφάσεις που πήρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μήπως το 2020 θα έχουμε έλλειψη πιστώσεων. Γιατί η περσινή μας τροπολογία, κύριε Μουρεσάν, ε, ε, υπέστη περικοπή, βεβαίως, πρόεδρε στην συνδιαλλαγή, καθώς ε, συμφωνούσαμε τον προϋπολογισμό για το 2018, αποφασίσαμε να αυξήσουμε τα ποσά και βάσει των οσο μαθαιναμε μαθαίναμε από πολλά κράτη-μέλη, αλλά και εν ώψη ε, ε, της ακόμα υψηλής ανεργίας των νέων. Και πραγματικά θέλουμε να δούμε να θα απορροφηθούν αυτά τα κονδύλια θα δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι σε περίπτωση που χρειαστούν περισσότερα ε, θα αντιδράσει. Θα δούμε και φέτος τη συνδιαλλαγή τι θα γίνει όταν θα αποφασίσουμε τα ποσά, κύριε Πρόεδρε, για το 19. Αλλά από πλευρά μου, σαφέστατα το πρόβλημα της ανεργίας των νέων δεν έχει λυθεί ακόμα και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ε, ότι θα έχει ε, αρκετή πρικοδότηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει τη λειτουργία του προγράμματο Αυτό μπορεί να μην ευθύνει τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού αλλά άλλων γενικών διευθύνσεων, αλλά εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το, πρόβλημα, το πρόγραμμα εφαρμόζεται σωστά και ανταποκρίνεται στην αποστολή. Très bien. Eh bien, je crois que nous allons pouvoir en Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα το αφήσουμε εδώ αυτό το θέμα τώρα των πληρωμών. Ευχαριστώ τον κύριο Ρέλ για την παρουσία του και θα ε, όσα μας είπε πολύ συγκεκριμένα στην αλλαγή αυτή απόψε. Και θα δώσω έλεγα το λόγο στο Jens Geier για να μας μιλήσει για το επόμενο θέμα. Και αφορά ε, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Κοινωνικό Ταμείο το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ήδη... Ε, ε, είχαμε κάνει μια ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό ήδη. Για να σας δώσω μια εικόνα, το τρέχον πολίτης δημοσιονομικό πλαίσιο δεν ε, έχει ικανοποιήσει το Ευρωκοινοβούλιο. Μας έδωσε ηρεμιστικά το Συμβούλιο όμως. Ε, ήταν αυτές, αυτά κάποια χρηματοδοτικά ε, μέσα γιατί η Επιτροπή είχε περιορισμένα ε, χρηματοδοτικά μέσα άλλα ηρεμιστικά ήταν ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε χρήματα από τα διευθυντικά ταμεία με την προπτική ότι αυτό το παθηματικό θα πρέπει τα αποθηματικά επιδόσεων να κάνουν αρκετά, να πράξουν αρκετά τα κράτη-μέλη και θα μιλήσουμε τώρα για αυτά τα παθηματικά επίδοσης. Αποφάσισε τελικά να μην τα θέσει στη διάθεση για τον στόχο αυτό, αλλά να δοκιμάσει αν αυτά τα παθηματικά επίδοση μπορούν να χρησιμοποιηθούν με προτάσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η υπεύθυνη επιτροπή, η αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής και είναι πολύ ξεκάθαρη στάση της. Όλες οι ομάδες προτείνουν να μην αλλάξει αυτή η πρόταση επιτροπής, απλά να την απορρίψουμε. Το παρακολουθώ αυτό το φάκελο και στις υπόλοιπες επιτροπές. Στην Ήτρε ισχύει το ίδιο. Και αυτή είναι και η πρόταση που κάνω και σε αυτή την επιτροπή. Προσωπικά και ίσως διαφοροποιούμε από κάποιους μέσα στην ομάδα μου, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα αν τα τα ταμεία σε σχέση με τους στόχους να κατανοηθούν σε συγκεκριμένα προγράμματα στα κρατημέλη. Αν πρώτον υπάρξει ομοφωνία, συμφωνηρώ με τα κρατημέλη, το, η αρχή της επικουρικότητας είναι πολύ σημαντική εδώ και δεύτερον αν θα επίσης ε, έχω επιφυλάξεις ε, για συμφωνίες σαν αυτές που γίνονται το 2013 να υπάρξουν αλλαγές στην πορεία γιατί θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη βασίζονται σε αυτά τα κονδύλια και θα έπρεπε να αλλάξει η στοχοθέτηση και το τελευταίο επιχείρημα μου είναι ένα πιο χειροπιαστό η Επιτροπή εξετάζει την εκπλήρωση των παραμέτρων τι θα κάνει όμως το 2019 το μόνο που μπορώ να φανταστώ δεν ξέρω τι μπορεί να μας εξηγήσει ο κύριος Αυτό που μπορώ να προβλέψω είναι ότι τα διευθυντικά ταμεία θα έχουν καθυστερήσεις και το 2019 θα πρέπει να εξετάσουμε θα είμαστε στο πρώτο τελευταίο τόσο ε, του τρέχοντος πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου και σύμφωνα με το νη 1 μπορούμε για τα επόμενα δύο χρόνια να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια και δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουμε ε, ουσιαστικά για τις προτεραιότητες στα κράτη-μέλη. Θεωρώ ότι δεν θα μπορούσαμε να το πράξουμε αυτό. Άλλη παρατήρηση που έχει να κάνει επί της αρχής έχουμε μια καλή ιδέα εδώ σε αυτήν την Επιτροπή και ξέρουμε ποιες είναι αντιδράσει στα υπόλοιπα όργανα. Υπάρχουν εκεί, θα προκύψουν νομικά θέματα ενδεχομένω. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, γιατί πρέπει ε, να έχουμε, να αντιμετωπίσουμε άλλα όργανα στη λήψη των αποφάσεων για μια ουσιαστικά ρύθμιση την οποία δεν την θέλαμε ποτέ. Και γι' αυτό ε, η πρόταση μου είναι να την απορρίψουμε την πρόταση αυτή. Voilà, donc proposition de... Πρόταση απόρριψη ε, από πλευρά του εισηγητού. Ποιο θέλει το λόγο, ο κύριο Φερνάντε. Από του κύριου εισηγητέ, δεν βλέπω κανέναν μεταξύ των παρόντων συναδέλφων. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φερνάντης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να επαναλάβω κάτι που είπα την περασμένη φορά που ανταλλάξαμε απόψεις για το συγκεκριμένο θέμα και την κατάσταση. Εγώ κατανοώ τα επιχειρήματα εκείνων που είναι αντίθετοι και επιθυμούν την απόρριψη. Διότι θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει προηγούμενο, γιατί το αποθεματικό επίδοσης είχε σχεδιαστεί για τα προγράμματα που δούλευαν καλύτερα και όχι για το σκοπό που έχουμε τώρα. Από την άλλη όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Δεν είναι υποχρεωτικό για τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτό το αποθεματικό επίδοσης για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε κάθε χώρα δεν είναι υποχρεωτικό. Θα πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε αυτό. Διότι αν δίνουμε στα κράτη-μέλη μια επιπλέον δυνατότητα να χρησιμοποιούν χρήματα που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, αυτό σημαίνει περισσότερη ευελιξία. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να ζητάμε ευελιξία. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα και έχω την τάση να συμφωνήσω με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα πρέπει όμως να το συζητήσουμε. Γιατί έχουμε άλλη μία δυνατότητα. Είναι ένα συν, ένα επιπλέον ατού που έχουμε στα χέρια μας. Να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν ένα αποθεματικό σε εθελοντική βάση και όχι υποχρεωτικά. Ε, ξέρω εγώ. Αν το δεχόμαστε όμως, παρόλο που βλέπω να απορρίπτεται, αυτό δεν θα μπορούσε καμία περίπτωση να αποτελέσει προηγούμενο. Και τα χρήματα για τα τα ταμεία είναι ένα πράγμα και τα χρήματα για το Ταμείο Συνοχής είναι άλλο πράγμα, διαφορετικό. Και αν γίνουν οι διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις, τα κονδύλια από την πολιτική συνοχής μπορεί να έχουν μια επιπλέον συνεισφορά και επιτυχία. Και η εκτέλεση του προϋπολογισμού μπορεί να είναι και πιο αποτελεσματική και να βοηθήσει για να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα και καλύτερα. Χρόνο έχουμε ακόμα για τη συζήτηση αυτή. Δεν ξέρω πώς το δικαιολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τις αμφιβολίες που ακούμε και που σας ανέπτυξα εδώ. Αλλά επιμένω, εάν αρμόδια επιτροπή επί της ουσίας έχει άλλα επιχειρήματα, η Ρέτζη, θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Αλλά εκείνη είναι αρμόδια επί της ουσίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεπχέ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην παρούσα φάση δεν θέλω να ασχοληθώ με θέμα ουσίας, αλλά να πω ότι στην δική μου πολιτική ομάδα υπάρχουν ε, πάρα πολλές διαφορετικές θέσεις. Κάποιοι συμφωνούν με τον κύριο Γκάια και κάποιοι άλλοι συμφωνούν με την θεωρία την οποία ε, παρέθεσε ο κύριος Φερνάντες. Μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα μπορούσε να μας βοηθήσει λίγο στη συζήτηση που γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έχει ζητηθεί από τα κράτη-μέλη, υπάρχει ζήτηση από τα κράτη-μέλη για μια τέτοια πρόταση. Είναι μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα ρύθμιση ή στην παρούσα φάση υπάρχουν ακριβώς κράτη-μέλη τα οποία μας λέγουν ότι μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε ε, το αποθεματικό. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το λάβουμε υπόψη μας Δεν θα συμφωνήσουν όλοι μαζί μου φυσικά και δεν απαιτώ να γίνει κάτι τέτοιο. Πριν δώσω το λόγο θα δώσω στην Επιτροπή, θα το δώσω στην Γουάρδια Ζαμπάλ. Ευχαριστώ όπως και ο κάθε ένας από εμά έχει διαφορετικά στοιχεία και δεν θα χαθούμε στα επιμέρους στοιχεία. Νομίζω όμως ότι δεν υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στις θέσεις του κυρίου Γκάγερ ε, και του κυρίου Φερνάνδης. Νομίζω ότι αυτό ε, που έχουμε πάντα πει είναι ότι αν θέλετε ένα νέο πρόγραμμα, οκ, αλλά θα πρέπει να υπάρξει επιπλέον χρήμα στον προϋπολογισμό και δεν θα πρέπει να θυγούν συμφωνίες περίπλοκες όπως ε, για το ε, κοινωνικό ταμείο ή κάποιες συμφωνίες που έχουν γίνει για τους λεγόμενους καλούς μαθητές. Ε, τώρα αν υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσει μια προπαρασκευαστική, μια πιλωτική δράση για μεταρρυθμίσεις, ε, αυτό είναι άλλο θέμα, αυτό δεν θα πρέπει να γίνει με χρήματα τα οποία έχουν προβλεφθεί για άλλους στόχους. Θα δούμε λοιπόν σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα. Όπως και να έχουν τα πράγματα σε επίπεδο προϋπολογισμών θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στην πρακτική μας μέχρι σήμερα. Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα, πρέπει να βρεθούν νέα χρήματα και δεν θα πρέπει να μειώνονται άλλου είδους προγράμματα. Και νομίζω ότι δεν έχουμε διαφορετική άποψη από τον κύριο Φερνάντες, αλλά, βέβαια, Φερνάντες, αλλά δεν ξέρω μήπως δεν κατάλαβα καλά αυτά που έπαιρνε. Κύριε Ιουχέλα, Σας ζητήθηκαν κάποιες διευκρινήσεις από πλευράς του κυρίου Ντεπρέ. Τα κράτη-μέλη ε, εκφράζουν ε, ακριβώς αυτό που θα ονομάναμε μια κάποια ζήτηση ή στην ουσία είναι μια πρωτοβουλία δική σας με βάση τη δική σας εμπειρογνωμοσύνη. Για την ερώτηση του κυρίου Ντεπρέ θα πρέπει να ε, ενημερωθώ και θα σας γράψω μια γραπτή απάντηση. Θα σας στείλω μια γραπτή απάντηση. Καλώς ε, κύριε Ισηγητά για να κλείσουμε το θέμα αυτό. Δεν ακούσατε κάποια αντιεπιχειρήματα. Γκάια. Είναι γενικά ένα θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να οδηγήσει εύκολα σε μια κάποια συνένεση θα μπορούσα να απαντήσω σε εξή ε, την ερώτηση του κυρίου Ντεπρέ. Εξ όσων γνωρίζω εγώ, βέβαια δεν έχω, το έχω ψάξει σε μεγάλο βάθος, υπάρχει ένα κράτος μέλος που βλέπει θετικά αυτή την ιδέα και αυτή είναι η Πορτογαλία. Με σοσιαλιστική κυβέρνηση, λέει ο κύριος ε, ε, Φερνάντες. Ναι, ναι, όντως, λέει ο κύριος Γκάιερ. Ε, ο καθένας μπορεί να έχει τις δικές του απόψεις. Και το δείχνω ε, ε, εγώ αυτή τη στιγμή γιατί δεν συμφωνώ με μια σοσιαλιστική κυβέρνηση. Εσύ κάνεις ό,τι θέλεις. Λείπει Ζωζέ Μανουέλ, αγαπητέ Ζωζέ Μανουέλ. Για ιδεολογικού λόγου το κάνει εσύ όμω. Εν πάση περιπτώσει, είτε κυβερνούν σοσιαλδημοκράτε είτε όχι στην Πορτογαλία, ε, δεν υπάρχει και μαζική πίεση των κρατών μελών που έχουν τρέξει να την αγκαλιάσουν. Τι φοβερή ιδέα είχατε ας την υλοποιήσουμε και να την ε, χρησιμοποιήσουμε για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν, αλλά το θεωρώ αυτό ε, ένα πείραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δηλαδή αυτή η ιδέα να παίρνουμε χρήματα από τα τα ταμεία και να τα συνδέουμε με το ευρωπαϊκό εξάμεινο ή στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν μου αρέσει. Στο επόμενο PDP, αν θέλετε να το συζητήσουμε, δεν είμαι τελείως αντίθετος με την ιδέα αυτή. Ε, είμαι μάλλον στη μειοψηφία της ομάδας μου. Αλλά εκεί που διαπιστώθηκαν ελλείμματα, πιστεύω ότι μπορούν να βοηθήσουν ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά θα το συνέδεμε με ορισμένους όρους και προϋποθέσεις. Δηλαδή συμφωνία του κράτους μέλους και να δούμε και το σύνολο των κονδυλίων που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην δημιουργήσουμε τετελεσμένα έτσι εμπαρόδο. Αυτά. Εγώ είμαι υπέρ της απόρριψης. Ευχαριστώ. Αν θέλετε να κάνετε τροπολογία. Μπορείτε να το κάνετε. Το αργότερο όμως την 5η 12 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Να θυμίσω ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών θα γίνει στις 29 και 30 Αυγούστου και επί της ουσίας στην Περιφερειακή Επιτροπή την 9η Οκτωβρίου. Για τον κύριο Ντεμπρέ, ο οποίος ε, ε, φοράει... Α, έφυγε ο κύριος Ντεμπρέ. Σας ευχαριστώ. Τώρα, δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Κοινωνικός πυλώνας, ο κύριος Γκάιερ πάλι. Αναφερθήκατε σήμερα ακροθυγώς σε αυτό όταν υποδεχθήκαμε τους εκπροσώπους των εξωτερικών υπηρεσιών. Και πάλι ευχαριστώ. Αυξάνονται οι υπηρεσίες, οι οργανισμοί μεγάλη αύξηση με ένα νέο οργανισμό, την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, Απασχόλησης. Καταφέραμε αυτό το χρόνο, όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, να έχουμε μια θετική απόφαση από κοινού. Μαζί με το Συμβουλίο την Απόσπαση των Εργαζομένων να συμφωνήσουμε σε μια οδηγία, την, το στενισμό των ε, ε, υποδομών, των πόρων. Για να τα εγγυηθούμε όλα αυτά, προτείνει η Επιτροπή την δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας, ενός νέου οργανισμού η δομή δεν θα αλλάξει. Είναι μια νέα ε, υπηρεσία για να δυσφαλίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οι αρμοδιότητες στην ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας από την πλευρά μου δεν είναι επαρκή για να γίνει επιτυχής ε, εφαρμογή και θα πρότεινα να έχουμε βελτιώσεις ώστε να γίνει μια πιο αποδοτική εφαρμογή και αυτό θα γίνει με γνωμοδότηση budget 52 δισεκατομμυρίων ε, ευρώ εκατομμυρίων ευρώ θα έχει 40 εργαζόμενους, 140 εργαζόμενους. Και προκύπτει το ερώτημα εδώ, πώς θα χρηματοδοτήσουμε αυτόν τον ε, οργανισμό. Η κατευθυντήρια γραμμή θα έπρεπε να είναι, κατά την άποψή μου, εφόσον θα είναι φορέας προγραμμάτων που θα τρέχουν, θα είχε νόημα αυτά τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας να μεταφερθούν γιατί δεν υπάρχει διαφορά απόψεων για το αν θα ε, χρηματοδοτηθούν από την υπηρεσία αυτή από την Επιτροπή τα επιχειρησιακά προγράμματα και τα έξοδα. Ε, και για τη χρηματοδότησή τους, τη εκεί θα ήμουν πολύ προσεκτικός και δεν είμαι πεπισμένος ότι η πρόταση επιτροπή είναι σωστή να αφορά το 70% του προπολογισμού να προέρχεται από το πρόγραμμα ε, κοινωνικής ε, καινοτομίας θεωρώ ότι θα έχουμε χαμηλότερες επιδόσεις και θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί καλύτερα η αρχή και γι' αυτό κάνω την πρόταση στην Επιτροπή για τον οργανισμό αυτό να κάνουμε κάτι που έχουμε κάτι ήδη για άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα και τη εργασία. Να υπάρχει δηλαδή μια διοικητική ε, δομή που θα είναι τριμερής. Να υπάρχουν μέλη από ο, εργαζόμενους εργοδότες ώστε να εκπροσωπούνται όλα τα συμφέροντα. Merci. Ευχαριστώ κύριε Σίγητα. Ε, Γιάννης. Κάια, Ποιος θέλει το λόγο. Αυτός ο κύριος Αλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησής του για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Βασικές αρχές του ποινών κοινωνικών δικαιωμάτων, Ε, είναι ε, πολύ σημαντική η κοινωνική διάσταση και η διάσταση της εργασίας και η δίκαιη μετακίνηση των εργαζομένων. Χαιρετίζουμε λοιπόν αυτά ε, τα στοιχεία αλλά και την πρόταση του εισηγητή. Μια προσέγγιση με στόχο την αποτελεσματικότητα και την ξεκονόμηση πόρων. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 10 και 18 και το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε το Eurofund, το και ε, άλλες ε, δομές και αυτή είναι η σωστή προσέγγιση και υποστηρίζουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο να υπάρχει και ένα μέλος από την οργάνωση των ε, εργοδοτών και ένα μέλος από την συνδικάτα των εργαζομένων και ένα μέλος που να ορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, θα είναι πάνω από 80 τα μέλη όμως αν είναι ένας από κάθε κράτος, εργοδότης, εργοζόμενος κτλ. Όμως ε, ο καθένας θα έχει 11 υπαλλήλους. Στο Eurofound αυτοί οι 11 ε, εκπροσωπούν κυβερνήσεις, εργαζόμενους, εργοδότες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ έχουμε διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν. Αυτά τα γραφεία θα αναφέρονται στο πρώτο τμήμα ή και στο αντίστοιχο άρθρο. Δεύτερον, σε περίπτωση της Eurofound αναφέρονται ως μέλη του Προεδρείου ε, και οι δύο εκπρόσωποι που ορίζει η Κομισιόν. Θα πρέπει να ισχύσει το ίδιο και για τους εκπροσώπους ε, που ορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, μετά, πάντα στο άρθρο 18, στην παράγραφο 3, ε, γίνεται λόγος για το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπούν τα κράτη-μέλη και τα μέλη που εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να είναι συνεκτικά όλα αυτά με την πρόταση μας στην τροπολογία 10, νομίζω ότι θα πρέπει να προσθέσουμε και κάποιους όρους ε, για την εκπροσώπηση εργοδοτών εργαζομένων, καθώς επίσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου. Και τέλος, κάτι που δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά νομίζω αξίζει να υποθεί και να διευκρινιστεί, στη περίπτωση των παλιών οργανισμών, ε, τι γίνεται, γιατί με τη νέα ε, Στη νέα αρχή γίνεται λόγος για managing board το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ στις προηγούμενες δομές ήταν διαφορετική η ορολογία. Όχι ότι έχει μεγάλη σημασία, αλλά θέλω να το πω γι' αυτό. Ευχαριστώ. Um, thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να αρχίσω με μια παρατήρηση για το μάτς ε, το βράδυ. Και οι δύο εθνικές ομάδες έχουν βελτιώσει ε, το ποδόσφαιρό τους γιατί οι παίκτες τους παίζουν στο αγγλικό πρωτάθλημα που, που είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό και το καλύτερο στην Ευρώπη. Βέβαια αυτό αφορά το αυριανό μάτς, θα δούμε τι θα γίνει. Ε, καλωσορίζω πάρα πολύ την πρόταση αυτή ε, για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Είναι ε, πολύ καλή πρωτοβουλία και έπρεπε να έχει έρθει εδώ και καιρό, όπως και οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων αν υπήρχε τέτοιο πλαίσιο για να αντιμετωπίζει τις πρακτικές ε, ε, κάποιων ασυνείδητων εργοδοτών και ε, αυτών που προχωρούν σε καταχρήσεις, δεν ξέρω αν θα χρειαζόμαστε τέτοια αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση από 28 θα έχει 27 μέλη προσεχώς, αλλά καλή οργά παραποτέ, εν πάση Αυτή η αρχή θα πρέπει να έχει και κάποια πυγμή και κάποιες δυνατότητες να επεμβαίνει, να επιθεωρεί, να συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές, έτσι ώστε να φέρνει καλές ε, πρακτικές και βελτιώσεις και να εξαλείφει τις καταχρήσεις. Γιατί εάν αποτύχει, τότε θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση που θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη απογοήτευση από τη δυνατότητα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των ε, κρατών μελών με τους θεσμούς τους να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες του κανονικού κόσμου, των κανονικών φυσιολογικών ανθρώπων στην καθημερινή τους λειτουργία. Εκεί λοιπόν θα κρυθούμε. Το θέμα δεν είναι τα 50 εκατομμύρια ο προπολογισμό και θα πιάσει τόπο, αλλά εάν θα βελτιώσει την καθημερινότητα ε, των πολιτών. Βεβαίως θα χρειαστούν κάποια χρόνια, αλλά εάν δεν έχει αποτελέσματα πραγματικά τότε θα είναι πεταμένα λεφτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Όλμπριχτ. Uh, Έχω μια ερώτηση γιατί στην Επιτροπή, Επιτροπή δεν είναι μόνο σημαντικό για εμάς το θέμα των αστερικών στόχων, αλλά το πόσο θα κοστίσει και για το μελλοντικό πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Αν δούμε τα νούμερα που προτείνει η Επιτροπή, η Επιτροπή προτείνει να ανέβουμε με τις δαπάνες για τις, ε, τους οργανισμούς 700 εκατομμύρια πιο πάνω, αλλά, άρα αυτά είναι ακριβώς τα χρήματα που απαιτούνται γι' αυτό είναι εν για, αυτή για αυτόν τον οργανισμό και για άλλους οργανισμούς. Θα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό πρωτού συζητήσουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να είμαστε καλά ενημερωμένοι για το κόστος στα επερχόμενα έτη. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε την απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Πρόεδρος, κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι, καθυστέρησα πέντε λεπτά γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό το σημείο στη μέσα διαταξή. Αρχή λέει αυτό το πράγμα, είναι στα, στα αγγλικά είναι αρχή, authority. Είχαμε μέχρι τώρα οι BOAs, Institutions, Bodies, Offices, Agencies, οργανισμοί, φορείς, θεσμοί και δεν συμμαζεύεται. Γιατί δεν το λέτε οργανισμό, αφού είναι οργανισμός, γιατί το λέτε authority, αρχή. Και αυτό θα ε, μας διευκόλυνε πάρα πολύ τη ζωή και ε, το δημοσιονομικό κανονισμό και όλα τα έγγραφα αν είχαμε το θάρρος να το ονομάσουμε οργανισμό. Και το οργανόγραμμα και η σύνθεση και τα πάντα δείχνουν ότι είναι οργανισμός, αλλά δεν το λέμε οργανισμό. Για ποιο λόγο. Δεύτερη ερώτηση. Τι θα κάνει λοιπόν αυτή η authority τώρα η αρχή βλέπουμε επικαλύψεις άλλων οργανισμών αποκεντρωμένων ε, που λειτουργούν μέχρι τώρα. Και επίσης έχουμε και ένα συμβουλευτικό ρόλο. Και γι' αυτό το λόγο ε, ρωτώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξετάσει για αν αυτές οι νέες αρμοδιότητες που δεν είναι και τρομακτικά πολλές δεν, μπορούν, δεν θα μπορούσαν να ανατεθούν σε ένα ήδη υφιστάμενο οργανισμό δεν είναι πάρα πολύ σκόπιμο να δημιουργούμε συνέχεια νέους θεσμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 50 εκατομμύρια το 2024. Αυτά είναι λεφτά που θα πονέσουν γιατί θα μας λείψουν από αλλού. Μήπως έχει έρθει η ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας μοιήσει και μας ε, στις διάφορες σκέψεις της και προθέσεις της. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φερνάντες τελευταίος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλώ εξ ονόματος του κυρίου Πέτερ Σαβαρμά, ο οποίος ε, δυστυχώς ε, απουσιάζει και ζήτησε συγγνώμη για την αποσία του. Είναι σκιώδη συγγετής του ΕΛΚ για το θέμα αυτό. Ε, ευχαριστεί τον εισηγητή για τη δουλειά του και συμφωνεί με όλα σχεδόν, αλλά διαφωνεί ο κύριος Σαβαρμά πάντα, όχι εγώ, ε, ως προς την χρηματοδότηση. Διότι θεωρεί ότι θα πρέπει η χρηματοδότηση να γίνεται κυρίως ε, από μεταφορές πιστώσεων. Το άλλο αφορά την ε, τροπολογία 7 για το dumping το μισθολογικό. Και ο κύριος Σαβαρμά θεωρεί εκεί ότι δεν θα πρέπει η αρχή αυτή να ε, κάνει έρευνες και να αναλύει αυτή η authority αρχή να αναλύει τα θέματα του μισολογικού dumping. Ε, κάτι άλλο έχει να κάνει με την τροπολογία 8 και πάλι εκεί ο κύριος Σαβαρμά θεωρεί ότι η διαδικασία για τις παραβάσεις δεν έχει τη δέουσα μορφή και την κατάλληλη για να επιλύονται αυτά τα ζητήματα. Άλλο που λέει ο κύριος Βαρμά, τι γίνεται με το προϋπολογισμό βάση επιδόσεων και με τις συνέργειες μεταξύ διαφόρων θεσμών, ε, φορέων, αρχών και οργανισμών και πώς μπορεί αυτή να ενισχυθεί. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ουρέλη για να απαντήσει στις ερωτήσεις που έγιναν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να πω ότι εμένα δεν με πειράζει αυτή η αρχή εργασίας να ρίξει μια ματιά και στην κατάσταση απασχόλησης στα διάφορα κράτη-μέλη και αναρωτηθεί αν είναι ε, φυσιολογικό σε μια χώρα με πλήρη απασχόληση να έρχονται τόσο πολλοί εργαζομένοι εκτός της Ευρώπης και να διατηρούνται πάρα πολύ χαμηλοί μισθοί έτσι και να μην είναι υπέρ της ε, ε, προοδευτικής σύγκλησης των αποδοχών. Παρακαλώ, κύριε Ουρέλ, έχετε το λόγο. Ε, thank you, Chair. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το ερώτημα που ρώτησε του κύριου Ουλμπριχτ στην Επιτροπή, έχει σχέση με τον δημοσιονομικό αντίκτυπο για το επόμενο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο αντίκτυπος που αντικατοπτρίζεται στην ε, νομοθετική δήλωση υπερβαίνει το 2020, άρα φάρει και το επόμενο πολιτές πλαίσιο. Όλο αυτό έχει ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή στις προτάσεις της, όπως υποβλήθηκαν στις 2 Μαΐου και στις επόμενες εβδομάδες η Επιτροπή θα θέσει στη διάθεση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου ένα, μια αναλυτική κατάσταση για, όλες τις για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς σύμφωνα με την πρόταση της Δευτέρας Μαΐου. Αν το λάβετε αυτό το έργο, θα μπορείτε να δείτε και μόνοι σας αναλυτικά ε, τα δύο ερωτήματα από την κυρία Γκρέσλε. Γιατί δεν το ονομάζουμε οργανισμό agency και το ονομάζουμε αρχή. Δεν είναι η πρώτη υπηρεσία που ονομάζεται αρχή. Υπάρχει και η τραπεζική αρχή και άλλες οπτικές αρχές. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, θα προτιμούσα να σας απαντήσω εγγράφως. Όσον αφορά το άλλο ερώτημα, θεωρώ ότι χρειάζεται μια πιο σε βάθος απάντηση. Όσον αφορά τις επικαλύψεις με άλλες υπηρεσίες, θα επανέλθω και στα δύο σας ερωτήματα γραπτός. Ευχαριστώ. Κύριε Σιγητά, έχουμε πίεση χρόνου εξαιρετική. Λοιπόν, πάρα πολύ σύντομα σας παρακαλώ το συμπέρασμά σας. Δεν μπορεί να είμαι και εγώ πάρα πολύ σύντομος, διότι βασικά οι παρατηρήσεις του Πέτρη Σάβαρμα ήταν τέτοιες που δεν είναι. Ε, μόνο εκεί έχουμε κάποια μεγάλη διαφορά. Ε, είναι εποπτική αυτή η αρχή και ο οργανισμός και με κάθε σεβασμό απέναντι στο συνάδελφο Σαβαρμά πρέπει να πω το εξής αν αυτός ο οργανισμός είναι εποπτικός, χρειάζεται να έχει και δόντια, όπως λέμε στα γερμανικά. Και πώς εκφράζεται αυτό το πρόβλημα συχνά με αποσπασμένους εργαζομένους. Ήταν το μισθολογικό dumping. Οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται στη Γερμανία και πληρώνονται πολύ κάτω του νόμιμου μισθού ή τους πληρώνουν το κανονικό μισθό, αλλά τους αφαιρούν το κόστος στέγασης, για παράδειγμα. Και αν προτείνω στον κανονισμό να συμπεριληφθεί αυτό το μισθολογικό dumping, αυτό έχει να κάνει με παραβιάσεις ενδεχόμενες ε, της ε, οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων. Μπορεί, λέω, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Και αν θέλουμε πραγματικά να έχει πυγμή και δόντια μια τέτοια αρχή ή οργανισμός, θα πρέπει να προτείνουμε ότι όταν υπάρχει παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, το οποίο διαπιστώνει αυτή η αρχή, θα πρέπει να δρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέπε να προσφεύγει επί παραβάση στο δικαστήριο. Και με το συμπάθειο, άμα ε, θέλει κάποιος να είναι ισχυρή αυτή η αρχή δεν θα πρέπει να υιοθετήσει αυτά που λέει ο Σαβαρμά. Οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο 13 Φεβρουαρίου τη 12η μεσημβρινή. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει 29 και 30 Αυγούστου και στις 18 θα γίνει η συζήτηση επί της ουσίας. Για να ωφεληθούμε από την διερμηνία ας ψηφίσουμε λοιπόν αυτό που δεν ψηφίσαμε το πρωί. Ζητώ από το Γενικό Εισηγητή να μου πει αν πήρε τις ε, λεπτομέρειες τις οποίες περίμενε σχετικά με τη μεταφορά 18. Όχι, δεν πήρα καμία επιπλέον πληροφορία από το πρωί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήρθε σε επαφή μαζί μου, αλλά είναι παρούσα εδώ και θα ήθελα να σας ζητήσω να τους δώσουμε το λόγο, κύριε Πρόεδρε, για να δούμε αν υπάρχουν κάποιες διευκρινήσεις. Κύριε Ουρέλ, Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να επανέλθω και να αντιμετωπίσω με λεπτομερέστερο τρόπο τις ερωτήσεις τις οποίες έκανε η κυρία Γκρέσλε σήμερα το πρωί. Το σύνολο των πόρων για το καταπίστευμα για την Αφρική είναι 3,4 δις. Τα κράτη-μέλη έχουν συνεισφέρει 430 ε, εκατομμύρια. Οι πιο σημαντικές ε, συνεισφορές είναι από τη Γερμανία 157, η Ιταλία 110 και μετά όλες οι υπόλοιπες χώρες οι οποίες είναι αρκετά μικρότερες. Η Ολλανδία είναι τρίτη με 26 εκατομμύρια. Το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο έχει δώσει λοιπόν κάτι λιγότερο από 3 δις και ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός 666 εκατομμύρια σε επίπεδο εφαρμογής. Η Λειτουργική Επιτροπή του Καταπιστεύματος ενέκρινε για την Λίμνη Τσάδ και το σαχέλο 85 προγράμματα Συνολικά, όπως λέει η γραπτή μας απάντηση, 1 δις 466 εκατομμύρια. Αν προσθέσουμε σε αυτά το κόστος διαχείρισης, τότε φτάνουμε σε ένα συνολικό ποσό για 1,6 δις. Αυτό σημαίνει ότι έχει καταναλωθεί ουσιαστικά το σύνολο του διαθεσίμου το οποίο είχαμε διαθέσει στην περιοχή Σαχέλ και Τσάδ, λίμνη Τσάδ. Ένα δις 630 εκατομμύρια είχαμε προβλέψει και γι' αυτό α, εξηγούνται τα 27 διαθέσιμα εκατομμύρια. Οι διαφορές ανάμεσα στους πόρους λοιπόν που ήσαν διαθέσιμοι και στα ποσά τα οποία ήδη έχουν καταναλωθεί είναι 27 εκατομμύρια. Συνεπώς αυτή είναι η εξήγηση, αν και το ποσό στη μεταφορά είναι πάρα πολύ περιορισμένη, θα βοηθήσει να καλυφθούν κάποιες άμεσες ανάγκες οι οποίες έχουν εντοπιστεί. Σχετικά με το χρηματοδοτικό κενό, υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό για το σύνολο του καταπιστεύματος κατά 1,1 δις. Είπαμε λοιπόν στην απάντησή μας ότι 0,6 δις συνδέεται με την περιοχή Σαχέλ Λίμνη τσαρ Για να μπορέσουμε να κλείσουμε το κενό αυτό, ε, η μεταφορά αυτή θα καλύψει μόνο ένα πάρα πολύ μεγάλο τμήμα αυτού του μεγάλου χρηματοδοτικού κενού, είναι σαφές. Και αυτό το οποίο τώρα είπε το Συμβούλιο πριν δύο εβδομάδες, είναι ότι για να κλείσει εν μέρη το κενό, 500 εκατομμύρια θα γίνουν διαθέσιμα από το αποθεματικό του Αναπτυξιακού Ταμείου στο καταπίστευμα. Η απόφαση αυτή έγινε δεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα, την 6η Ιουλίου, και εξετάζεται από την Επιτροπή του Αναπτυξιακού μέσω της γραπτής διαδικασίας με τελική ε, ημερομηνία την επόμενη εβδομάδα. Αυτό θα μειώσει λοιπόν το 1,1 που μας λείπει δεν ξέρουμε ακριβώς θα δώσουμε στο Σαχέλ και τι ποσό θα δώσουμε στο Κέρας. Είναι κάτι που πρέπει να αποφασιστεί. Το Συμβούλιο ταυτόχρονα δεν έχει αποφασίσει ακόμα, αλλά έχει προσκαλέσει τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν περαιτέρω στο καταπίστευμα για την Αφρική, έτσι ώστε να κλείσει το υπόλοιπο κενό και έτσι το συνολικό 1,1 εκατομμύριο να καλυφθεί. Δεν έχουν αναλυφθεί επίσημα υποχρεώσεις από τα κράτη-μέλη ως προς αυτό. Μένει να γίνει αυτό. Μετά από τα 500, τη μεταφορά των 500 εκατομμυρίων, το κενό για το καταπίστευμα στο σύνολο θα είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια. Ελπίζω η απάντηση αυτή να σας καλύπτει. Ευχαριστώ. Σας καλύπτει, κύριε Γενική Εισηγητά. Πρόεδρε, δεδομένου του πεδίου εφαρμογής αυτής της μεταφοράς, είναι επαρκής αυτές οι εξηγήσει. Τώρα επικρατεί μεγαλύτερη σαφήνεια για το συγκεκριμένο, για το γενικότερο, όχι ακόμα, νομίζω μπορούμε να τα ψηφίσουμε. Alors, je Πολύ ωραία. Με ηλεκτρονική λοιπόν ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία και ψηφίζουμε. Όχι. Α, να πω ότι καλό θα ήταν οι μεγάλες ε, διακηρύξεις που ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, καλό θα ήταν να συνοδεύονται και από πράξεις, γιατί είναι τέτοια η διάσταση και το χάσμα που χωρίζει που μας προκαλούν από τρόποι μου και αγανάκτηση. Άρχεται η ψηφοφορία. Tout le monde a il Ψηφίσατε όλοι. Όχι. Ένας. Ακόμα πέρασε. Τις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 12 ψήφοι υπέρ και μία ψήφος κατά. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Λεβαντόφσκι, θα ήθελα να σας πω ότι λυπούμε για το γεγονός ότι η Προεδρία τη στιγμή που αναλαμβάνει η Αυστρία την Προεδρία του Συμβουλίου δεν θεώρησε σκόπιμο να έρθει ενώπιον της Επιτροπής Προϋπολογισμών να πήγε σε όλες τις υπόλοιπες επιτροπές. Εγώ τους είχα απευθύνει επιστολή μήπως δεν πήρανε το γράμμα γιατί ούτε απάντηση πήρα. Ήθελα να σας ε, απευθύνω αυτή τη λύπη μου και να τη μοιραστώ μαζί σας. Ο κύριος Λεβαντόφσκι τώρα για το Ταμείο Λεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, Ελλάδα, Λιθουανία και Πολωνία. Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Ε, αντίδραση ρουτίνας είναι αυτή. Ε, του Ταμείου Αλληλεγγύης ε, αλλά τα θέματα που καλύπτει δεν είναι καθόλου θέματα ρουτίνας γιατί είναι φυσικές καταστροφές και θεομηνίες. Τον Οκτώβριο του 2017 η Ελλάδα ε, ζήτησε μετά τους σεισμούς βοήθεια σε, μια, σε ένα νησί και σε κάποιες άλλες περιφέρειες. Αργότερα η Πολωνία μετά από καταστροφικές καταιγίδες και πλημμύρες στη δική μου ο περιοχή του Δεκέμβριο του 17 η Λιθουανία μετά τις ε, πλημμύρες και τον ε, Ιανουάριο του 18 ακολούθησε η Βουλγαρία μετά από τις πλημμύρες. Εδώ θα σταματήσει η διερμηνία σύμφωνα με την προηγούμενη ανακοίνωση καθότι σήμερα δεν παραχωρούμε υπέρβαση ωραρίου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας